επηρεάσουν αρνητικά την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα λίγη αυτή η συζήτηση. Επόμενο σημείο η έκθεση του Γεωργίου Τσίτσεστερ δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών. For the floor. Έχει λοιπόν το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζω αυτή την έκθεση που αναφέρει τα πεπραγμένα της Επιτροπής Αναφορών το 11. 998 αναφορές ελήφθησαν, λίγες απορρίφθηκαν, 550 και η στατιστική αυτή ανάλυση αναφέρεται ήδη από την αιτιολογική έκθεση γιατί είναι ενδιαφέροντα τα στοιχεία που περιέχει δηλαδή η προέλευση των αναφορών τα θέματα καθώς και οι χώρες από που οι χώρες των αναφερόντων. Τα πιο ενδιαφέροντα για αυτούς θέματα ήταν τα θεμελιώδη δικαιώματα, η εσωτερική αγορά και είναι επίσης ενδιαφέρον ότι οι περισσότεροι πολίτες μιας μεμονωμένης χώρας που κατέθεσαν αναφορές ήταν η Γερμανία και μετά η Ισπανία και η Ιταλία. Ενώ οι χώρες τις οποίες αφορούν τα θέματα είναι η Ισπανία και η Γερμανία με διαφορετική σειρά χώρες. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον διότι και οι επιστολές που λαμβάνω εγώ από τους εκλογείς μου δείχνουν ότι η χώρα μου που είναι έκτη ή έβδομη στον αριθμό ετούντων δείχνει ότι ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν οι Βρετανοί πολίτες την Ένωση δεν είναι εκείνος που θα αναμέναμε ή θα αναμέναμε πολύ περισσότερες αναφορές. Θα σας πω τώρα μερικά από τα θέματα που αναφέρει η έκθεσή μου. Πρώτον, το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών στην απόκτηση κατοικίας και οι ανησυχίες τους για το τι θα γινόταν με τις κατοικίες αυτές ε, ε, εάν αγόραζαν κατοικία σε άλλη χώρα μάλλον. 51 αναφορές έρχονταν από Ισπανούς δεν αφορούσαν ξένους που αγοράζουν εξοχικές κατοικίες, αλλά κατοικίες Ισπανών και αυτό το θέμα αναφέρθηκε πολλές φορές πέρυσι. Επίσης υπάρχει αυξανόμενος αριθμός αναφορών που θέτουν θέματα που δεν είναι δικαιοδοσία της Ένωσης. Ίσως αυτό να το θεωρήσουμε υπέρ ως θετικό δηλαδή ότι στρέφονται οι πολίτες σε εμά για να αναζητήσουν λύσεις. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, μεγάλος αριθμός πολιτών θέτουν θέματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς ε, με την ιστοσελίδα μας θελήσαμε να δημιουργήσουμε ένα ακριβώς πιο προσβάσιμο βήμα για τους πολίτες και χαιρετίζουμε τη συνεργασία που είχαμε με τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητή. Επαναλαμβάνουμε δε την υποστήριξή μας στο έργο του για την ταύτιση της κακοδιαχείρισης από ευρωπαϊκά όργανα. Θεωρούμε ότι η σωστή εφαρμογή της οδηγίας waste ή μάλλον της διαχείρισης των, των αποβλήτων είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό ιδίως αν το σχετίσουμε και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ακτές, στις ακτές της Ισπανίας που είναι θέμα που συνεχίζει να ενδιαφέρει τους πολίτες εκεί. Θέλω δύο λεπτά παραπάνω στο τέλος κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Τσίτσεστερ. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση. Ε, δίνω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Σεύκοβιτς και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Τσίτσεστερ ως εισηγητή επίσης την κυρία Ματσόνη και όλη την Επιτροπή Αναφορών της οποία η δράση αντικατοπτρίζεται στην έκθεση. Η έκθεση αναφέρεται στα πιο κοινά ε, θέματα που απασχολούν τους πολίτες στο, στο τομέα του περιβάλλοντος και των θεμελιών δικαιωμάτων. Το Κομισιόν και το Κοινοβούλιο συνεργάζονται στενά και θα συνεχίσουν να τα, ανταλλάσσουν πληροφορίες για αυτά τα θέματα. Η σημερινή συζήτηση είναι μια καλή ευκαιρία να υπογραμμίσω το πόσο ε, χαίρομαι για την δράση σας ε, στην, ε, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του άρθρου 227 της συνθήκης που επιτρέπει στους ε, πολίτες ε, ή και νομικά πρόσωπα να υποβάλουν αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Κομισιόν είναι ιδιαίτερα χαρούμενη που μπορεί να συνεισφέρει στην εργασία σας. για μας αποτελεί σημαντική επένδυση ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά το αξίζει γιατί με αυτόν τον τρόπο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Η συνεργασία μας δείχνει ότι είμαστε προσιλωμένοι στο να θέτουμε τους πολίτες μπροστά ε, πάνω απ' όλα. Όπως αναφέρεται πολύ σωστά και στην έκθεση Λίχτεμπεργκ που θα συζητηθεί αμέσως μετά, σήμερα το βράδυ, η Επιτροπή Αναφορών παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο ο σύνδεσμος ανάμεσα στους πολίτες ε, το κοινό και αφενός και την Κομισιόν από την άλλη. Γι' αυτό το λόγο περιμένουμε ε, κάθε χρόνο με ανυπομονησία την έκθεση για την εφαρμογή του κοινοτικού νόμου. Ε, στην επόμενη ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του της κοινωτικής νομοθεσίας που υιοθετηθεί τις επόμενες εβδομάδες ε, σκοπεύουμε να ε, αναφέρουμε τον αριθμό των ε, περιπτώσεων που ξεκίνησαν από την Επιτροπή Αναφορών. με αυτά τα στο μυαλό να επαναλάβω ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σας και με την Επιτροπή Αναφορών όπως η έκθεση Τσίτσεστερ αναφέρει μας ζητάτε, για, ζητάτε τη βοήθειά μας για πάνω από το 50% των άνω των χιλίων ε, τιμάτων αναφορών που ε, λάβατε το προηγούμενο έτος. Ε, α, παρακολουθούμε και την εξέλιξη όλων των ε, αναφορών που φτάνουν σε εμά και ε, περιμένουμε ότι θα συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία και στο μέλλον. Αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια για, την, για τις πρωτοβουλίες ε, ε, Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών. Από την 1η Απριλίου ένα νέο εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας βρίσκεται στα χέρια των πολιτών μας που είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Τα αρχικά τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν έχουν πλέον επιληθεί η Κομισιόν έχει θέσει τους δικούς της σερβερς στην υπηρεσία των πολιτών βοηθώντας τους ε, για την διαδικασία πιστοποίησης των υπογραφών. Τρεις ε, πρωτοβουλίες ε, έχουν ήδη ξεκινήσει και συλλέγουν πλέον υπογραφές online αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά έχω δεσμευθεί οι πολίτες να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν 100% αυτό το νέο τους δικαίωμα. Και θα ήθελα επίση να υπογραμμίσω ότι η Κομισιόν αναμένει να συνεχίσει και να βελτιώσει τη συνεργασία της με την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Τώρα ο κύριος Πρέδα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ξέρετε η Επιτροπή Αναφορών δεν ε, είναι θέμα που συζητιέται συχνά στην Ολομέλεια. Παρ' όλα αυτά η εργασία της είναι πάρα πολύ σημαντική. Δέχεται τα παράπονα των πολιτών και γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι προασπίζει τα δικαιώματά τους. Γι' αυτόν τον λόγο η Επιτροπή Αναφορών οργανώνει πολλές ακροάσεις κάθε χρόνο και ε, διατηρεί σταθερό διάλογο με την Κομισιόν, με αρχές των χωρών μελών και με άλλα όργανα όπως τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Δυστυχώς οι μισές περίπου αναφορές που κατατίθενται δεν είναι αποδεκτές διότι τα θέματά τους είναι εκτός των δικαιοδοσιών της Ένωσης. Πρέπει λοιπόν στο μέλλον να γίνει μια καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ειδικότερα η Επιτροπή Αναφορών θα έπρεπε να οργανώσει ακροάσεις και για το θέμα της ε, πρωτοβουλίας των πολιτών που ανέφερε και ο Επίτροπος για να βελτιωθεί έτσι η πληροφόρηση. Επίσης, εκτός από τις χώρες που ανέφερε ο κύριος Τσίτσεστερ, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία ως χώρες που κατέθεσαν τις περισσότερες αναφορές, Μετά έρχεται η Πολωνία και η Ρουμανία έρχονται στην τέταρτη και πέμπτη θέση. Άρα και οι παλαιές και οι νέες χώρες μέλη ενδιαφέρονται για την προάσπιση των ενδιαφέρονται οι πολίτες για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους όπως και για την προστασία του περιβάλλοντος και της εσωτερικής αγοράς. Και αυτό δεν είναι τυχαίο γιατί είναι τα σημαντικότερα θέματα της ενωσιακής ζωής. Τελειώνω λέγοντας ότι θα πρέπει να στηρίξουμε την Επιτροπή Αναφορών που είναι ένα εργαλείο διαλόγου μεταξύ του Κοινοβουλίου και των πολιτών. Και τώρα για 1,5 λεπτό ο κύριος Μποστινάρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ε, συγχαρώ τον ε, εισηγητή κύριο Τσίτσεστερ για την πολύ καλή έκθεση και για την εξαιρετική ε, συνεργασία κατά την κατάρτιση αυτής της εκθέσεως διότι είχαμε πάρα πολλές αναφορές στον προηγούμενο χρόνο σχετικά με την νομοθεσία στα θέματα του περιβάλλοντος και θα ήθελα να να τονίσω αυτό το χαρακτηριστικό διότι αναφέρεται στην ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών και την διαφύλαξη των θησαυρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό υπενθυμίζω στον Επίτροπο Ποτόσνικ την οδηγία που αναφέρεται, με τον, στον ε, έλεγχο της ανεκτικότητος και θα παρακολουθήσω η αναμόρφωση αυτής της οδηγίας να βασιστεί σε σαφή κριτήρια εξασφαλίζοντας την ουδετερότητα και την αντικειμενικότητα ε, των ε, μελετών που θα ε, αξιολογήσουν τις επιπτώσεις διότι οι Ευρωπαίοι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να εκφράσουν μέσω της Επιτροπής μας τις ανησυχίες τους ε, και γι' αυτό παρακαλώ τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει την ελεύθερη διακίνηση όλων των Ευρωπαίων πολιτών ασχέτως της φυλής. Ευχαριστώ. Τώρα για δύο λεπτά η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι από τις πλέον σημαντικές διότι διασυνδέει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με τους πολίτες και εγώ έχω ορισμένου αριθμούς και βλέπουμε το 1997 ε, είχαμε 20.000 ε, αναφορές ε, και ε, ε, ε, τώρα είδαμε ότι η Επιτροπή μας ασχολήθηκε πολύ σοβαρά με 323 αναφορές πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι ασχολούμαστε εις βάθος με το θέμα όπως ελέγχθη πολύ σημαντικό είναι το περιβάλλον διότι πρέπει να αξιολογήσουμε όπως άλλωστε αναφέρθηκε και ε, την οδηγία για την ε, εφαρμογή και τις ε, περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις. Έχουμε αντιμετωπίσει πολλές περιπτώσεις όπου υπήρξαν αρνητικές επιπτώσεις και σε μια δικιά μου περιοχή την Καρνεκάρα. Ένα άλλο σύστημα το οποίο μας έχει απασχολήσει είναι οι δυσχέρειες και δυσκολίες για την ελεύθερη διακίνηση ιδίω για άτομα που χρειάζεται να συνοδεύονται από έναν προσωπικό βοηθό και ε, η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών ακόμη δεν είναι ικανοποιητική ε, μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Και τέλος ε, πρέπει να τονίσω ένα, μια άλλη διαπίστωση την οποία έκανα στην Επιτροπή. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, ειλικρινείς, να προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε την κατάσταση και να μην ε, τσουλάμε τις ευθύνε σε κάποιον άλλον. Και τώρα η κυρία Άουκεν για τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να προσθέσω και εγώ τη φωνή μου σε αυτήν των συναδέλφων που ευχαρίστησαν τον κύριο Τσίτσεστερ. Δεν θα επαναλάβω τα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Ε, συνοπτικά όμως ε, να πω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η Επιτροπή Αναφορών ε, θα πρωταγωνιστήσει στα τεκτενόμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο μέλλον και θα τη χρησιμοποιούν οι πολίτες. Ένα θέμα θέλω να τονίσω είναι ο νόμος περί παράκτηων περιοχών της Ισπανίας. Τώρα στην παράγραφο 18 αναφέρεται ότι ε, κράζετε μάλλον τη χαρά σας για την ισπανική συνεργασία της συνεργασίας της Ισπανίας. Ε, δεν φαντάζομαι να το εννοείτε. Το ε, νομοσχέδιο αυτό πέρασε πολύ βιαστικά από το, από το Κοινοβούλιο Ισπανίας και ελπίζω αύριο θα υποστηρίξετε την τροπολογία μας υπαρθμών 5 και την υπαρθμών 6 ε, ε, που αναφέρει ότι ο νόμος περί παράκτιων ζωνών της Ισπανίας ε, παραβαίνει το, έρχεται σε αντίθεση με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2009. Δεν είναι δυνατόν να, να υπερασπίσουμε τις ακτές και την φύση ε, δίνοντας περισσότερα δικαιώματα στους ε, ιδιοκτήτες κατοικιών εκεί. Ε, δεν θέλουμε να δώσουμε ωφέλη στις, σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες πράγμα το οποίο υπάρχει κίνδυνος να γίνει μέσω εκ των υστέρων και αναδρομικής τακτοποίησης και νομιμοποίησης αυθαιρέτων. Λοιπόν, πολλά είναι τα καλά της έκθεσής σας. Ελπίζω όμως ότι ε, θα εξασφαλίσουμε πλειοψηφία και για την, τον, ε, την πρότασή μας να στείλουμε ένα μήνυμα προς την Ισπανία. Ε, δεν θα τελειώσουμε τι εργασίε μα ε, ε, πριν ε, τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος, ο ισπανικό νόμο. Γι' αυτό λόγο είναι ευκαιρία αύριο να δώσουμε μήνυμα προ την Ισπανία. Χρησιμοποιείται η έκθεση Αουκεν για να νομιμοποιηθεί δήθεν το νομοσχέδιο αυτό που θα εξετάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να στείλουμε μήνυμα προς την Ισπανία ότι δεν είναι δυνατόν να αγνοούν το Κοινοβούλιο και την έκθεση Άουκεν ε, του 2009. Ευχαριστώ. Thank you very much. And just now... Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στον κύριο Τσαρνιέτσικη για τρία λεπτά. Ε- Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του, του Τσεχικού Κοινοβουλίου έχει κάνει σχετικές δηλώσεις αλλά ας επανέλθω στο θέμα μας. Η σημασία της Επιτροπής Αναφορών είναι πολύ μεγάλη γιατί είναι η τελευταία προσφυγή η τελευταία ευκαιρία που έχουν μερικοί πολίτες για να προσφύγουν στην Ένωση, να υποβάλουν τα, παράπονό τα παράπονά τους. Και δεν έχουν άλλη πρόσβαση παρά μέσω αυτής της Επιτροπής Αναφορών. Και οι προηγούμενοι ανέφεραν τη σημασία της με συγκεκριμένα παραδείγματα. Η Επιτροπή αυτή αναφορών χειρίζεται πάρα πολύ σημαντικά πολιτικός θέματα. Και κατά την προηγούμενη θητεία Παραδείγματο χάρη ασχολήθηκε με το θέμα του North Stream του αεριαγωγού της Βαλτικής Δυστυχώς όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε εγκρίνει τελικά μία γνωμοδότηση, μία, αναψήφισμα που αντετάχθη στην αρνητική θέση των περισσότερων χωρών μελών γι' αυτό. Η Ισπανία, θα συμπενθυμίζω ότι είχε το θέμα του καταλανικού ραδιοφώνου ΚΟΠΕ και οι αρχές είχαν αρνηθεί την άδεια της λειτουργίας του. Ενώ η Επιτροπή Αναφορών έκανε έναν αγώνα σε συνεργασία με τον πρόεδρο του Καταναλικού Κοινοβουλίου ή εναντίον του πρόεδρου του Καταναλικού Κοινοβουλίου και ο αγώνας αυτός κερδίθηκε. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει αποτέλεσμα η εργασία της Επιτροπής αυτής. Θυμηθείτε και την πολωνική εκείνη περίπτωση όπου ένας πολίτης είχε προσφύγει στην Επιτροπή Αναφορών για το θέμα των αυτοκινήτων ευκαιρίας που εισάγονταν στην Πολωνία και των δασμών που τους επιβάλλονταν. Να, τέτοια συγκεκριμένα παραδείγματα επιτυχιών είναι που χτίζουν τη φήμη της Ένωσης. Ευχαριστώ τώρα για 1,5 λεπτό ο κύριος Αλαβράκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος ε, Τσίτσεστερ εισπράττει συγχαρητήρια για την καλή εκθεσή του και παρακαλώ να προσθεθούν και τα δικά μου. Το έργο της Επιτροπής Αναφορών, κύριε Πρόεδρε, είναι εξαιρετικά σημαντικό για την προάσπιση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών και των δημοκρατικών θεσμών στον χώρο της Ευρώπης. Θετικά κρίνεται το γεγονός ότι ο αριθμός των νέων αναφορών που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή το 2011 αυξήθηκε. Η Επιτροπή ασχολήθηκε με ποικίλε αναφορές. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, η εσωτερική αγορά, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των πολιτών, καθώς και τα περιβαλλοντολογικά ζητήματα ήταν οι βασικοί τομείς που βρίσκονταν στο επίκεντρο των εργασιών της Επιτροπής. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, παρατηρείται αύξηση των αναφορών πάνω στον τομέα των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών υποθέσεων ως απόρρια της τρέχουσας κρίσης χρέους. Στο περιεχόμενο των αναφορών που έρχονται στην Επιτροπή κατοπτρίζεται η ανησυχία και τα θέματα που πλήττουν και απασχολούν τους Ευρωπαίους πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο σημαντική κρίνεται η έκκληση για βελτίωση της δικτυακής πύλης της επιτροπής μέσα από τον ιστότοπο του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα η διαφάνεια της διαδικασίας των αναφορών και η παροχή καλύτερης πληροφόρησης στους ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much. And just now for minutes, Mr. Ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Γιάρ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή κύριο Τσίτσεστερ για την εξαιρετική έκθεση η οποία προωθεί τις επιτυχίες της Επιτροπής αλλά θέτει και τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων και, και διευκρινεί τα σημεία που χρήζουν ακόμη βελτίωσης διότι πρέπει να προσφέρουμε στους πολίτες της Ευρώπης τη δυνατότητα να μπορούν να προσφύγουν εάν αισθάνονται ότι αδικούνται ή στην Ευρώπη και υπάρχει μια ευρία ποικιλία θεμάτων και έχουμε προσπαθήσει με θάρρος να αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα και να έχουμε άμεση επαφή με τους πολίτες αφενός και να τους συνδέσουμε με την Ευρωπαϊκή Ίνηση. Γι' αυτό και γίνονται ε, διάφορες αποστολές για την διαπίστωση στοιχείων για να μπορούν και οι πολίτες να έρθουν για πρώτη φορά σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό ακόμη είναι ένας καλός στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας. Βέβαια κάθε ε, ε, εργασία μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο και κατά τη γνώμη μου καταρχήν θα πρέπει να μειώσουμε το χρόνο επεξεργασίας, να μην ε, καθυστερούμε και ε, να μην καθυστερεί τόσο πολύ και η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία πολλές φορές περιμένει για πολύ χρόνο τα στοιχεία από τα κράτη-μέλη πρέπει να μπορέσουμε συγχρόνως να βελτιώσουμε τη συνεργασία με τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διότι πολλές από τις ε, αναφορές που λαμβάνουμε προωθούν συζητούνται στις επιτροφές και αυτό θα εμπλουτίσει την όλη διαδικασία. Ευχαριστώ κύριο Κάσμαν τώρα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ συγχαρητήρια στον κύριο Τσίτσεστερ για την εξαιρετική του έκθεση. Η Επιτροπή Αναφορών ε, είναι ο ενδιάμεσος ανάμεσα στους πολίτες ε, αφενός και τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη αφετέρου. Μερικές φορές το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν το σωστό. Και το ίδιο κάναμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε και σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της Ισπανίας. Όμως από το 2004 ε, ε, καμία από τις ισπανικές ε, αναφορές ε, ιδιοκτητών δεν επιλήθηκε θετικά οι πολλοί νόμοι μεταξύ αυτών και ο νόμος περί παρακτήρων ζωνών ε, αφαρμόζονται λανθασμένα και αυτό οδηγεί σε καταδαφίσεις κλπ. Ε, ελπίζω ότι ε, η επιτροπή που έχει δημιουργηθεί για να συζητήσει το ζήτημα από την Επιτροπή Αναφορών θα οδηγήσει σε πραγματικές πράξεις και όχι μόνο σε λόγια. Σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, η ομάδα των σοσιαλιστών έχει υποβάλει μια τροπολογία ε, η οποία αντικατοπτρίζει τη βασική αρχή μας, την ισότητα. Ε, οι οικογένειες ίδιου φύλου, οι οικογένειες Ρωμά κλπ. υποφέρουν ιδιαίτερως από περιορισμού στην ελευθερία κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχουμε δει πολλές φορές. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στα κράτη-μέλη ότι η οδηγία του 2004 38-2004 ε, τους επιβάλλει ε, να μην εφαρμόζουν διακρίσεις στην ε, υποδοχή ε, οποιονδήποτε διακινούμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Βοητσεκόφσκι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συγχαίρω και εγώ τον κύριο Τσίτσεστερ με πολύ καλή έκθεσή του. Να υπογραμμίσω επίσης τον ρόλο της Επιτροπής ε, Αναφορών και το έργο της που πολλές φορές επισκιάζεται από το έργο άλλων επιτροπών άλλων επιτροπών πολύ συχνά ασχολούνται με νομοθετικά κείμενα κλπ. Όμως η Επιτροπή Αναφορών έχει σημαντικό ρόλο επαφής με τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι και η αποστολή της, να γνωρίζουμε πώς λειτουργεί και πώς εφαρμόζεται το κοινωνικό δίκαιο στα κράτη-μέλη μέσα από περιπτώσεις συγκεκριμένων πολιτών ε, έτσι βλέπουμε το κατά πόσον ε, πιάνει τόπο το νομοθετικό μας έργο. Ε, υπάρχουν πολλοί βέβαια που αποστέλουν αναφορές ε, ε, τις οποίες θα πρέπει να εξετάσει η Κομισιόν. Η Κομισιόν είναι ουδέτερη. Ε, ε ίσως στο ε, μέλλον οι αναφορές θα πρέπει να εξετάζονται και από άλλες επιτροπές. Όχι μόνο από την Επιτροπή Αναφορών. Ε, ίσως λείπουν κάποιες πληροφορίες από αυτήν την έκθεση του κ. Τσίτσεστερ, για παράδειγμα ε, την αποτελεσματικότητα των αναφορών, τι τελικά αλλάζει χάρη σε, σε αυτές τις αναφορές. Αν καταφέρνουν να ε, λάβουν κάποια επανόρθωση οι πολίτες ε, που έχουν υποβάλει αναφορές. Και επίσης τι γίνεται με τις αναφορές οι οποίες δεν ήταν παραδεκτές. Ασφαλώς δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν όλες οι αναφορές μία προς μία, αλλά οι πολίτες οι οποίοι αποστέλουν αναφορές, ε, ιδιαίτερω αναφορές οι οποίες δεν μπορούν να εξεταστούν από το Κοινοβούλιο, αυτοί οι πολίτες θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να ικανοποιηθούν με μια απάντηση, για παράδειγμα ε, παραπέμποντας αυτές τις αναφορές ε, στις αρμόδιες αρχές του Α ή του Β κράτους μέλους. Αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο για τους πολίτες. Ε, θα μπορούσα επίσης να αναφέρω το θέμα του εναρμονισμένου ΦΠΑ το οποίο θα μπορούσε να εξετάσει η Επιτροπή Αναφορών στο μέλλον. Ξέρουμε ότι στην Πολωνία παράδειγμα υπάρχουν πολλά παράπονα εξαιτία του ότι το κοινοτικό δίκαιο δεν εφαρμόζεται ε, σωστά στην Πολωνία. Ευχαριστώ κύριε Ματσόνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σχετικά με τα θέματα τα οποία εξετάσαμε ε, δεν θα επαναλάβω αυτά που ήδη αναλύθησαν. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τσίτσεστερ για την εργασία του και τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις και μπορώ να σας πω ότι ο απολογισμός μπορεί να αποδειχθεί ε, επικοδομητικός σχετικά με τον αριθμό των αναφορών που, που υπευλήθησαν για αυτές που έγιναν παραδεκτές ή όχι. Υπάρχει μία σαφής βελτίωση των εργασιών της, της Επιτροπής μας και ε, των μέσων που τις διετέθησαν. Επίσης, ε, οι πρωτοβουλίες οι οποίες ξεκίνησαν για να βελτιωθεί η πρόσβαση των ε, πολιτών προς ε, την Επιτροπή μας ήταν πολύ σημαντικές ε, και απετέλεσαν μία προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι εκθέσεις σε αυτή την ομίγυρη αποδεικνύουν τη χρησιμότητα των κειμένων αυτών για τους πολίτες και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που ελήφθησαν. Η, η Επιτροπή Αναφορών άλλωστε έχει ε, αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες όπως άλλωστε το είπε και ο Επίτροπος ε, Σευκοβίτς και τον ευχαριστώ για την ε, προσοχή την οποία αναπέδωσε στο θέμα και βλέπουμε ότι υπάρχει ένας χαρακτήρας πιο δημοκρατικός στην ε, Επιτροπή Αναφορών ε, από το 2011 που συμβάλλει στην ε, οικοδόμηση της Ευρώπης των λαών. Ευχαριστώ που σεβαστήκατε τον χρόνο και τώρα για ένα λεπτό η κυρία Γκέριγκεν Έντενμπεργκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι πολύ ε, σημαντική η η Επιτροπή Αναφορών για να παρακολουθεί ε, την ε, εργασία τις εργασίες και τις αναφορές στο θέμα των πολιτών και τα βασικά, τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν ένα πολύ βασικό τομέα ε, εξού και βλέπουμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, στην τελευταία του απόφαση ε, τόνισε τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εδώ πρέπει να τονίσουμε την πρόθεση του One Stop Shop για την προώθηση και αυτή η παρακολούθηση πρέπει να συνεχιστεί. Θα πρέπει να συνεχιστεί, η εποπτεία θα πρέπει να ενταθεί, ιδίω όσον αφορά το περιβαλλοντολογικό δίκαιο για διάφορους τομές. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κέλλη να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επενήσω τον κύριο Τσέτσεστερ για την εξαιρετική του έκθεση και επίσης να συγχαρώ και τους άλλους συναδέλφους οι οποίοι συνεργάστηκαν. Το 2011 είδαμε ε, ότι έγινε ένας απολογισμός που απέδειξε ότι πάρα πολλές αναφορές είχαν πλέον τύχη επεξεργασίας που ασχολούντουσαν με πολλά θέματα και έχω την τιμή να παρουσιάσω μία αναφορά εν ονόματι των ψηφοφόρων της περιοχής μου και ε, επί έξι χρόνια δεν είχαν αποτέλεσμα. Δεν μπορούσαν να προωθήσουν την αναφορά τους, επρόκειτο για τοξικά απόβλητα και πήγαινε από τον Άννα στην Κοϊάφα η όλη υπόθεση, αλλά τέλος ε, υπήρξε ένα αποτέλεσμα ε, και είδαμε ότι ε, όταν διαπιστώθηκε 37% περισσότερο ποσοστό καρκίνων ε, ε, ήταν δυνατόν να ληφθεί μία απόφαση και δόθη διορία τριών μοιρών στην κυβέρνηση να καθαρίσει τον χώρο που είναι ένα πολύ επικοδομητικό παράδειγμα για το τι μπορεί να επιτύχει η Επιτροπή των Αναφορών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για ένα λεπτό κύριο Σταμπάτζη. Thank Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Επιτροπή Αναφορών είναι η συνείδηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Αποτελεί και μία σπίδα ε, για την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εξού και στηρίζω την έκθεση Τσίτσεστερ διότι θεωρώ ότι η, έκθεση, η Επιτροπή Αναφορών εκτελεί εξαιρετική εργασία και ουσιαστική και τυπική και υπάρχει θαυμάσια συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Επιτροπής Αναφορών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό διότι πρόκειται για θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία έχουν παραβιαστεί και είδαμε τον αριθμό των προσφάτων αναφορών από την Ουγγαρία επειδή αναδρομικά η Ουγγαρέζικη κυβέρνηση ε, τροποποίησε ε, τι ε, συντάξεις ε, των αστυνομικών οργάνων και θεωρώ ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο κύριος Βαλέσα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Το περασμένο έτος εστιάσαμε την δουλειά της Επιτροπής Αναφορών σε δύο θέματα κυρίως, προστασία του περιβάλλοντος και θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, αυτή τη χρονιά ο αριθμός των καταγγελιών ε, έφτασε στις 1416 ε, ένας αριθμός βέβαια ε, τέτοιων αυτών αναφορών δεν ήταν παραδεκτός θα πρέπει λοιπόν να πληροφορήσουμε καλύτερα τους πολίτες για το νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη λειτουργία της Επιτροπής η απόφαση του ε, Κοινοβουλίου ε, να συμπεριλάβει ε, και την, την Επιτροπή Αναφορών και στο, στις για το θέμα της, των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλίων Πολιτών ήταν πολύ θετική. Η Επιτροπή Αναφορών άλλωστε έχει πολλή εμπειρία στις σχέσεις με τους πολίτες, είναι ο ρόλος της θα είναι θετικός. Ε, είναι λοιπόν πολύ, σημαντική, οι, πολύ σημαντικές οι αποφάσεις για την βελτίωση ε, της επαφής με τους πολίτες, για παράδειγμα η βελτίωση της ε, σελίδας στο ίντερνετ. θα πρέπει επίσης να δημιουργηθεί και μια ε, μονοαπευθυντική θηρίδα για τους πολίτες. Ευχαριστώ. Κυρία Γκέντς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, θέλω να ευχαριστήσω για την εξαιρετική έκθεση η οποία αποδεικνύει πόσο σημαντική είναι η, ε, πόσο σημαντικός είναι ο σεβασμός των δικαιωμάτων και ότι πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν και να εξασκούν τα δικαιώματά τους ε, να θεωρούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν έγκυρο συνομιλητή και βλέπουμε από τον αριθμό των αναφορών πόσο αυστηρή ε, έχουν καταστεί οι ε, έλεγχοι σε εθνικό επίπεδο ε, γιατί βλέπουμε ότι ο αριθμός επέρασε από 26 131 και ε, ε, προσπαθούμε συγχρόνως να εξεύρουμε μία δίκαια λύση και αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε ένα πνεύμα συνεργασίας με τις Ευρωπαϊκές Επιτροπής και τις δικιάς μας Ο κύριος Μπουλάν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Επιτροπή Αναφορών αυτόματα συνδέθηκε με τις δραστηριότητες της πρωτοβουλίας των πολιτών. Για μένα είναι το κυριότερο θέμα, γιατί οι πολίτες ήδη είχαν μια επιτροπή όπου μπορούσαν να υποβάλουν παράπονά τους και τώρα μπορούν να υποβάλουν και προτάσεις για βελτίωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Γι' αυτό η Επιτροπή Αναφορών μπορεί να θεωρηθεί ως ο κυριότερος συνομιλητής του πολίτη και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματά της και τα ιστοποθετήσεις της συχνά οι πολίτες αντιμετωπίζουν νομικά προβλήματα και μπερδέματα. Α, τα προβλήματα μπορεί να είναι ευρωπαϊκά, αλλά για να είναι ευρωπαϊκές και οι λύσεις πρέπει να γίνει κάτι παραπάνω. Δεν έχουν συνδεθεί τα δύο θέματα, το πρόβλημα με τη λύση, δηλαδή σε ενουσιακό επίπεδο. Παραδείγματος χάρη ή τα διαζύγια μεταξύ δια... ανθρώπων διαφορετικής προέλευσης. Έχουν υποβληθεί αναφορές από τη Γερμανία. Υπάρχουν πολλοί μεικτοί γάμοι, αλλά τα κοινοβούλια δεν έχουν αντιδράσει ακόμη νομοθετικά. Για να έχουν το δικαίωμα όλοι οι πολίτες σε εθνικό διαμεσολαβητή, ιδιαίτερα στη Γερμανία που στέλνει πολλές αναφορές, όπως γίνεται Στη Γαλλία δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά κάτι τέτοιο. Ενώ δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τα προβλήματα σε ενωσιακό επίπεδο και οι λύσεις να είναι μόνο εθνικές. Έτσι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις, ε, σε αυτά που ζητάνε οι πολίτες. Χρειάζονται να διαθέσουμε περισσότερα μέσα στη δράση μας λοιπόν. Με συγχωρείτε αλλά πρέπει να τηρείτε το χρόνο σας. Το, γιατί μετά θα φύγουν οι διερμηνεύτριες. Λοιπόν, τώρα για 1,5 λεπτό η κυρία Μπασέσκου. Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή Αναφορών μπορεί να είναι η καλύτερη μέθοδος για να δημιουργηθεί ένας δημόσιος διάλογος για τα προβλήματα που αφορούν τον απλό πολίτη στα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινή του ζωή. Το 2011 η Επιτροπή Αναφορών ασχολήθηκε πολλές φορές με θέματα με σεβασμού θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αλλά απ' την άλλη πολύ μεγάλος αριθμός αναφορών αφορούν πολιτικά προβλήματα που είναι εθνικής δικαιοδοσίας και όχι ενωσιακής. Και γι' αυτό απορρίπτονται από την αρχή. Παράδειγμα, η ελευθεροτυπία, η, τα ορυχεία στη Ρώσια Μοντάνα στη Ρουμανία, τα δέσποτα σκυλιά ή το αέριο, το συστολιστικό αέριο. Τέτοιου είδους αναφορές θα έπρεπε να αναλύονται περισσότερο για να βλέπουμε αν πρόκειται για επίκαιρα πολιτικά προβλήματα σε μια χώρα μέλος ή όχι έγινε προσπάθεια πολιτικοποίησης της δραστηριότητας της Επιτροπής στη Ρουμανία και σε άλλες χώρες για συγκεκριμένα προβλήματα. Εμείς είμαστε ευρωβουλευτέ και ο καθένας ανήκει σε κάποιο κόμμα. Την Επιτροπή αυτή όμως τη χρησιμοποιούμε μόνο για τα συμφέρον, την εξυπηρέτηση των πολιτών και όχι των κομμάτων μας. Κανείς δεν έχει ζητήσει το λόγο στην οφθαλμοθυρία και γι' αυτό θα ακούσουμε αμέσως τον κύριο Επίτροπο Σευκόβιτς. Ορίστε κύριο Επίτροπέ μου. Θέλω να ευχαριστήσω μια ακόμα φορά τον κύριο Τσίτσεστερ, την Επιτροπή Αναφορών, την κυρία Ματσόνη για την εξαιρετική συνεργασία της Επιτροπής αυτής με την Κομισιόν θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, να διευρύνουμε τη συνεργασία μας και να δούμε πώς μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική. Γι' αυτό το λόγο στην ε, έκθεση του επόμενου έτους για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου θα συμπεριλάβουμε όπως είπα και στις αρχές μου παρατηρήσεις ε, το input της Επιτροπής Αναφορών αναφέροντας συγκεκριμένα ε, τον αριθμό των ε, αναφορών που έχουν ε, σχέση με την εφαρμογή του κοινωτικού δικαίου. Θα ήθελα να πω σε σχέση με την σημερινή συζήτηση ότι χαιρόμαστε που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σκοπεύει να αναβαθμίσει το διαδικτυατικό του τόπο συμπεριλαμβάνοντας και τις αντιδράσεις της ε, Κομισιόν στις αναφορές που φτάνουν στα χέρια μας. Εξαιρετική αυτή η πρωτοβουλία και σίγουρα θα συνεργαστούμε μαζί σας γι' αυτό. Επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο να αναφέρω, να σχολιάσω δύο μόνο θέματα. Ε, πρώτον, σε ό,τι αφορά τις αναφορές για θέματα περιβάλλοντος και στην ε, παρέμβαση που αφορούσε την αναθεώρηση ε, το, της οδηγίας για τις ε, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η πρωτοβουλία υιοθετήθηκε, η πρόταση υιοθετήθηκε στις 26 Οκτωβρίου. Ε, θα θέλαμε η διαδικασία υιοθέτηση τη να ε, γίνει. Ε, συγγνώμη, θέλουμε να καταστήσουμε την διαδικασία ε, των εκθέσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων πιο απλή, λιγότερο γραφειοκρατική και πιο αντικειμενική. Ε, νομίζω ότι ε, αυτό θα εξασφάλιζε περισσότερο τους ε, πολίτες και θα τους διαβεβαίωνε ότι αξιολογούνται σωστά όλες οι περιβαλλοντικές πτυχές. Σε ό,τι αφορά τώρα τον νόμο για τις παράκτητες ζώνες στην Ισπανία, στον οποίο αναφέρθηκε η κυρία Άουκεν και ο κύριος Κάσμαν, να σας πω ότι η Κομισιόν έχει θίξει το θέμα στις Ισπανικές Αρχές, επανειλημμένως μάλιστα τα τελευταία χρόνια ακριβώς διότι ε, γνωρίζουμε τον αριθμό των αναφορών που προέρχονται και από Ισπανούς πολίτες αλλά και γενικότερα από Ευρωπαίους πολίτες. Ε, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις του θέματος, ιδιαίτερα το καινούριο νομοσχέδιο το οποίο υποβλήθηκε στο Ισπανικό Κοινοβούλιο. Βρισκόμαστε σε επαφή με τις Ισπανικές Αρχές και η και η Κομισιόν θα, ακολουθήσει πολύ θα παρακολουθήσει πολύ προσεκτικά ε, το τι θα ε, ψηφίσει το Ισπανικό Κοινοβούλιο για να δει αν επηρεάζει την υπόλοιπη Ευρώπη ή όχι. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να δώσω τέλος το λόγο στον κύριο Τσίτσεστερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους για τα καλά τους λόγια. ένιωσα σαν να ήταν ένας φίλος μου που μου χάιδευε το αυτί και μου τα έλεγε. Ευχαριστώ όμως και όλους τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν στην ε, συγγραφή της έκθεσης αυτής με τόσο καλό πνεύμα συνεργασίας από την Επιτροπή Αναφορών αλλά και για την αναγνώριση της δουλειάς μας. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την Κομισιόν γιατί όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι και η Κομισιόν παίζει σημαντικό ρόλο στη διεκπαιρέωση των ετοιμάτων μας για αντίδραση στις αιτήσει αναφορές των πολιτών. Η έκθεση αυτή εντυπωσιάστηκα από τον αριθμό εξάλλου των μελών που ζήτησαν το λόγο δείχνει τη σημασία που δίνουν οι βουλευτές οι συνάδελφοι για τη δουλειά μας που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για να ακουστεί η φωνή των πολιτών. Ένα θέμα θέλω να σχολιάσω που ανέφερε η συνάδελφος κυρία Όκεν. Παραπονούμενη, λογικό και αυτό και θεμητό, ότι για το θέμα των Ισπανικών αρχών προσπαθώ να είμαι όσο ευγενέστερος γίνεται με τις Ισπανικές αρχές γιατί έχω πολίτες μου και στο Γιβραλτάρ αλλά η έκθεση γράφει